Άρχεται η συνεδρίαση. Άρχεται η συνεδρίαση. Κυρίες και κύριοι. Κολίγ Συνάδελφε Γιάτσεκ, παρακαλώ καθίστε. Ε, η κυρία Γκόμες θα ήθελε να λάβει το λόγο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας πω ότι παρουσίασαν οι κυρίες Ντέβα και Σιμάνσκι κάποιες τροπολογίες ε, για το θέμα των εκτρώσεων Εσείς... Ε, νομίζω ότι θα ήθελα να, υπάρχουν, να υπάρχει εξή προσθήκη. Θα ήθελα και για τα παιδιά κυρίως που ζουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως τα κορίτσια, να μην υπάρχουν διακρίσεις. Εγώ αυτό το οποίο προσπαθώ να κάνω είναι να μπορέσω να προστατεύσω τα κορίτσια ε, πριν να γεννηθούν κατά της επιλεκτικής έκστρωσης. Και βεβαίως αυτό δεν έχει να κάνει τίποτε με την διακοπή της κοίησης. Αυτό το οποίο προσπαθώ εγώ να κάνω είναι να προσπαθήσω να κάνω κάτι το ορθό. Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε οι συνάδελφοι που προανέφερα να δημιουργήσουν πρόβλημα χρησιμοποιώντας το δικό μου όνομα. Λοιπόν, εγώ θα ψηφίσω αυτές τις τρεις τροπολογίες των κυρίων Ντέβα Σιμάνσκι που αναφέρονται στο θέμα αυτό που προανέφερα. Ευχαριστώ. για τη δήλωση αυτή, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν θα ήθελα να ανακοινώσω ότι το βραβείο Σαχάροφ για το 2009 κατά τη διάσκεψη των Προέδρων σήμερα για το βραβείο Ζαχάροφ λοιπόν κατά τη διάσκεψη των Προέδρων σήμερα αποφασίστηκε ότι θα απονεμηθεί στην οργάνωση Memorial. Θα ήθελα λοιπόν Αλεγκάλγκο, Ψέργια Γκαβαλιόβ, Λουτμίλα Αλεξέγεβα είναι τα τρία ονόματα των μελών της οργάνωσης Memorial που εκπροσωπούν ε, την ε, μάλλον που αγωνίζονται για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εμείς με το βραβείο Ζαχάροφ, με την αποσνομή μάλλον του βραβείου Ζαχάροφ, συμβάλλουμε στο να εξαλειφθεί η, ο φόβος, η βία και άλλες μορφές διώξεων που ε, που χρησιμοποιούνται εναντίον των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να ασκήσουν τα δικαιώματά του, δικαιώματα όπω ελευθερία τη σκέψη, ελευθερία του λόγου και ελευθερία του γραπτού λόγου. Θα πρέπει να είμαστε όλοι ελεύθεροι, να ασκούμε ελεύθερα τα δικαιώματά μας, να διατυπώνουμε ελεύθερα τις σκέψεις μας, διότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μοιραζόμαστε και να γνωρίζουμε την αλήθεια. Και ήταν ε, ιδιαίτερο προνόμιο για μένα να κάνω αυτή την ανακοίνωση ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά επίσης και ως μέλος του κινήματος αλληλεγγύης, διότι και εμείς αντιμετωπίσαμε στο παρελθόν παρόμοια προβλήματα στην Πολωνία ε, παρόμοια με αυτά τα οποία αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας και οι εταίροι μας στην Ρωσική Ομοσπονδία. Και με μεγάλη ικανοποίηση μπορώ να δηλώσω ότι η αλήθεια και η ελευθερία τελικά ε, κυριαρχούν. Τούτο συνέβη σε πάρα πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και το γεγονός ότι το γεγονός ότι υπάρχουν Ρώσοι οι οποίοι αγωνίζονται για την αλήθεια και την ελευθερία ε, είναι πολύ ευχάριστο για την Ευρώπη αλλά και για τους υπερασπιστές των, βασικών δικαιωμάτων. Γι' αυτό λοιπόν υποστηρίζουμε τις ενέργειές τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, Τώρα ένα γενικό σχόλιο. Από το 1989, δηλαδή πάνω από 20 χρόνια, και ε, υπό το πνεύμα του Αντρέη Ζαχάροφ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απονέμει τα βραβεία Ζαχάροφ σε άτομα και οργανισμούς που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, σήμερα λοιπόν ε, ανατρέχουμε σε αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν κατά των διώξεων των ε, ε, εκτοπίσεων και άλλων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, σκεφτόμαστε αυτούς τους απλούς ανθρώπους οι οποίοι διακινδύνευσαν ακόμα και τη ζωή τους. Ε, το βραβείο αυτό λοιπόν απονέμεται σε άτομα αλλά και σε οργανώσεις που υπερασπίζονται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης και σε οργανώσεις γυναικών. Η ελευθερία της σκέψης είναι μια πανανθρώπινη αξία. Και θα ήθελα να τονίσω ότι οι υποψήφοι που δεν έλαβαν φέτος το βραβείο Ζαχάροφ, που ήταν όμως υποψήφοι για το βραβείο αυτό, επίσης θα έχουν την υποστήριξή μας και θα πρέπει να συνεχίσουμε να ομιλούμε και για αυτούς ως ανθρώπους τους οποίους θα θυμόμαστε, θα θυμόμαστε το έργο τους. Το γεγονός ότι τους ε, ε, περιελάβαμε στον κατάλογο των υποψηφίων σημαίνει ότι προσδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στο έργο και τις πράξεις τους. Όχι μόνο δηλαδή ο νικητής του βραβείου Ζαχάροφ αλλά και οι υποψήφοι αυτού του βραβείου θα πρέπει να τύχουν του σεβασμού μας. Η απονομή του βραβείου θα λάβει χώρα την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο. Και τώρα περνούμε στην ψηφοφορία του σχεδίου Γενικού Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010 και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Σούριαν που είναι ο εισηγητής. Έχετε το λόγο κύριε εισηγητά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.